Σε υποβάλλονται σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο θα θεωρείται ότι εγκρίνονται αν μέχρι 24 ώρες προθεσμίας από μια κοινοβουλευτική ομάδα ή από ευρωβουλευτές δεν δηλωθεί ότι ζητείται να τεθούν υποψήφιση. Είναι και στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης θα εμφαίνονται. Σαν επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κοινή συζήτηση για το θέμα της δικαιοσύνης.